Χότς και Κλωρόζοβσκι από 27 Νοεμβρίου 2015 και έρχονται να αντικαταστήσουν τον κύριο Κρόβατσικ και τον κύριο Γιατσικίεβιτς. Καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους και σύμφωνα με τον κανονισμό μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Σύμφωνα με τον κανονισμό μας έχουν πλήρη δικαιώματα και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου και